Όχι, υπάρχει διερμηνία, ναι βεβαίως. Ναι, ναι. Η διερμηνία λειτουργεί. Ο κύριος Γκάιερ μου είπε πως βεβαίως με καταλαβαίνει και χωρίς ε, διερμηνία. Αυτό είναι γιατί δεν μίλησα τη διάλεκτο βεβαίως ε, της ε, Σουηδίας. Λοιπόν, περνάμε στο δημόσιο μήμα τη συνεδρίας. Πρώτα απ' όλα να σα πω πω σε μυστική ψηφοφορία η Επιτροπή μας δέχτηκε την πρόταση τη βουλγαρική κυβέρνηση για την πλήρωση της θέσης στο ελεγκτικό συνέδριο από την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα κατά πλειοψηφία, με μεγάλη πλειοψηφία με 17 ψήφους υπέρ 5 κατά 2 κατά με και 5 αποχές συγχαίρω λοιπόν την κυρία Ιβάνοβα και Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω λοιπόν ξανά τον Επίτροπο, τον κύριο Σέμετα. Ξέρετε πως συνεργαζόμαστε στενά σε πολλούς τομείς. Χαιρόμαστε για το ότι βρίσκεται εδώ πέρα σήμερα για να δώσει απαντήσεις, όπως και σε άλλες ε, βεβαίως επιτροπές. Είναι και για μας σημαντικό να γνωρίζουμε το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν έτσι ώστε και εμείς οι αιρετοί, οι βουλευτές να μπορούμε να προγραμματίζουμε για το πώς θα συνεισφέρουμε και εμείς ε, στη δουλειά της Κομισιόν και βεβαίως ε, υπήρχαν και οι συζητήσεις στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να διατίθενται κονδύλια χωρίς απαλλαγή, οπότε ελπίζουμε η Κομισιόν να μας βοηθήσει εδώ πέρα όσον αφορά το ζήτημα της απαλλαγής έναντι του Συμβουλίου, κάτι το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και βεβαίως κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί επί σειρά ετών είναι η αποστολή των ετησίων εκθέσεων των κρατών μελών μετά από χρόνια που αναμέναμε μια τέτοια κίνηση βλέπουμε πως στην φετινή διαδικασία απαλλαγής ανακοίνωσε ο κύριος Σέμετα πως θα μας δώσουν αυτές τις ετήσιες συνόψεις οπότε τηρείται έστω και αργά η υπόσχεση αυτή των κρατών μελών και σας ευχαριστώ εδώ πέρα για το ότι στηρίξατε αυτή την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου κατά το οποίο ζητήσαμε επιμόνως και ελπίζω να λειτουργήσει το σύστημα. Λοιπόν, δεν θέλω να προκαταλάβω τη συζήτηση βεβαίω, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που μας απασχολούν. Θεωρώ πως έχουμε ένα κοινό ενδιαφέρον στους τομείς της ε, προστασίας ε, των οικονομικών συμφερόντων της ε, Ένωσης και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της κοινή διαχείρισης των μέσων, των κοντιλίων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης που βρίσκεται σε αυτή την κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται στον πολιτικό τριμερή διάλογο με Συμβούλιο και Κομισιόν και εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού πάντα θίγουμε αυτό το θέμα και θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα για το πώς εκτιμάει η Κομισιόν την ε, κατάσταση, τι σκοπεύετε να κάνετε για να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Σέμετα. Έχετε το λόγο. Ε, thank you for this. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Πριν αρχίσω την ε, παρουσία μου, θα ήθελα να σας αποδείξω ότι κρατώ τις υποσχέσεις μου. Έχω μαζί μου ένα πακέτο με αιτήσεις ε, συνόψεις με πληροφορίες ε, για τα κράτη-μέλη που δεν σας είχα δώσει μέχρι τώρα. Μαζί με την επιστολή του Γενικού Διευθυντή του Walter Defa της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειών με τους κανόνες ε, που διέπουν αυτές τις αιτήσει συνοπτικές εκθέσεις. Ορίστε με χαρά τη τις υποσχέσεις μου και σας παραδίδω. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας και για την ανταλλαγή απόψεων που αποτελεί ουσιώδες τμήμα του διαλόγου μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων εν ώψη του μελλοντικού προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ ευχαριστώ θα συζητήσω θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας. Τα θεσμικά μα όργανα συμμερίζονται του βασικού στόχου τη προάσπισης των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη εξασφάλιση ε, υγιού δημοσιονομική διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων με μηχανισμού που εξασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ε, που θα χρησιμοποιείται με νόμιμο και τακτικό τρόπο και θα αξιοποιείται από αυτούς που τη χρειάζονται και την δικαιούνται. Αυτή είναι ε, και αρχή όχι μόνο υγιούς νομικής διαχείρισης, αλλά αποτελεσματικότητας ε, δικαιοσύνης και ισοτιμίας. Το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012, που εθετήθηκε πέρσι τον Νοέμβριο, είχε στόχο να αντιμετωπίσει τις κατεπίγουσες ανάγκες που ανέκυψαν ε, εξαιτία της κρίσης. Από ό,τι ξέρουμε σήμερα, η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να είναι ευάλωτη και ποικίλει από χώρα σε χώρα. Γενικώ πάντως βρισκόμαστε σε ήπια ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στη συνέχεια σε σταθερό και σταθερή και υφόρο ανάπτυξη, όπως αναφέρεται στον οδικό μας χάρτη το Οκτωβρίου του 2011. Στο μήνυμά μας τη ημέρα Σούμαν απευθύναμε έκκληση σε όλους τους φορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντείνουν τις προσπάθειές τους ε, για μεγέθυνση και απασχόληση επιταχύνονται στην εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε συγκεκριμένες συστάσεις προκειμένου να γίνει μεταρρύθμιση των αναγκών και να δημιουργηθούν νέες ε, θέσεις ευκαιρίας, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να ανοίξει το μέσο των υπηρεσιών ε, και των δικτύων. Επίσης προτείναμε ένα προϋπολογισμό που προωθεί την ανάπτυξη για το 2013 και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 υπό αυτό το πρίσμα επίσης. Γνωρίζουμε ότι τα δημόσια οικονομικά υφίστανται τεράστιες πιέσεις και μάλιστα στους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι δημόσιοι φορείς να εισπράττουν σωστά τα χρήματα και να τα αξιοποιούν με αποτελεσματικό τρόπο. Ε, να δούμε τα έσοδα πρώτα. Η σωστή ίσπραξη ε, των εσόδων είναι θεμελιώδους σημασία. Είναι ένας τομέας που θα πρέπει να είναι διαφανής και αποτελεσματικός και οι μηχανισμοί του το ίδιο. Θα επικεντρωθώ σε δύο βασικές προτεραιότητες στον τομέα αυτό. Ίσπραξη του ΦΠΑ και ίσπραξη των έμεσων φόρων κατανάλωσης. Ήδη το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κατήρτισε μια συντονισμένη στρατηγική για να βελτιώσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε επικοδομητικέ συζητήσει με τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Τώρα είμαστε σε θέση να πούμε ότι σχεδόν όλε οι νομοθετικέ προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για το θέμα αυτό της φοροαποφυγή του ΦΠΑ έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί από τα κράτη-μέλη. Ως δεύτερο βήμα θα πρέπει να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των μέτρων αυτών. Αλλά θα πρέπει να γίνουν και διάφορα άλλα πράγματα. Μετά την διαδικασία αξιολόγησης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κρίνει κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσει ή αν υπάρχουν κάποιε αδυναμίε μετά την πλήρη εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία. Συμπληρωματικά, μάλιστα, μέτρα πρόκειται να συνοδεύσουν αυτή τη διαδικασία παρακολούθηση και ελέγχου. Για παράδειγμα, θα διερευνήσουμε την δυνατότητα θέσπιση ε, ενό πανευρωπαϊκού επιτελείου ε, ανάλυση διασυνοριακού κινδύνου με εμπειρογνώμονε από τις Εθνικές φορολογικέ Αρχές προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί ο πολυμερής έλεγχος. Αυτή τη στιγμή μάλιστα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποιους μηχανισμούς αντίδρασης και να αποφύγουμε απάτη τύπου καρουσέλ με πολύ άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας στις αγωγές, δηλαδή την διαδικασία υπαριθμό 42 όπως είναι γνωστή, σας διαβεβαιώ ότι οι Γενικέ Διευθύνσει Προπολογισμού και τα ΞΟΥΝΤ έχουν διενεργήσει ελέγχου σε όλα τα κράτη-μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στα κράτη-μέλη που πλήττονται από τι μεγαλύτερε αδυναμίε στη διαδικασία αυτή. ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη στρατηγική, την ελληνική στρατηγική για τη διαχείριση του κινδύνου. Και μάλιστα έγιναν αξιολογήσει πριν την μεταρρύθμιση οδηγία για το ΦΠΑ και πριν την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων από τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξετάζει την ε, αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και πρόκειται να αναλάβει κατάλληλη δράση και να υποβάλει προτάσεις ακόμη και αναθεώρησης της νομοθεσίας αν παραστεί ανάγκη. Σε ό,τι αφορά του ειδικού φόρου κατανάλωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα πρόγραμμα εργασία κατά του λαθρεμπορίου σιγαρέτων και υνοπνευματοδοποτών ποτών στα ανατολικά σύνορα τον Ιούλιο του 2011. Γιατί το λαθρεμπόριο σιγαρέτων οδηγεί σε απώλειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τα ε, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Ως εκ τούτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί θεμελιώδη την πάταξη αυτού του λαθρεμπορίου σιγαρέτων. Και μάλιστα η ΟΛΑΦ ε, διενεργεί ε, έρευνες για διεθνές λαθρεμπόριο σιγαρέτων και επίσης συντονίζει διάφορες τέτοιες ε, διώξεις στα κράτη-μέλη και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη έχει κοινέ τελωνιακές επιχειρήσεις όπου κατέληξαν σε κατάσχεση μεγάλων αριθμών ε, λαθρέων σιγαρέτων τα τελευταία χρόνια. Επαναλαμβάνω τη δέσμευσή μου υπέρ της εφαρμογής αυτού του σχεδίου δράσης και θα εθαρρύνω τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΟΛΑΦ προκειμένου να περιοριστεί αισθητά το λαθρεμπόριο σιγαρέτων στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα τον έλεγχο των ιδίων πόρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τη δράση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την ίσπραξη τελωνιακών δασμών. Με βάση τα ετήσια προγράμματα ε, αξιολόγηση των κινδύνων, πραγματοποιεί δειγματοληπτικού ελέγχου στα κράτη-μέλη, προκειμένου να ελέγξει τι ε, πρακτικέ και διαδικασίε του σε ό,τι αφορά τη θέσπιση, το λογιστικό έλεγχο και την ανάκτηση ε, ιδίων πόρων. Και μάλιστα φέτος έγιναν πάρα από 30 έλεγχοι, τα πορίσματα των οποίων ε, ε, δεν μένουν χωρίς συνέχεια. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη γίνεται μια παρακολούθηση μέχρι το να ληφθεί δράση. Περίπου 76 εκατομμύρια ευρώ ζητήθηκαν από τα κράτη-μέλη πέρυσι εξαιτία των οικονομικών τους ευθύνων. Σε ό,τι αφορά τι δαπάνε τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για την εκτέλεση του κοινοτικού προπολογισμού και τη διαχείριση των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων. Θα λάβετε μάλιστα ως ονούπο μία συνοπτική έκθεση των, ε, του Συλλογικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ανάληψη συλλογικής ευθύνης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλιστα η απόφαση αυτή θα στηριχθεί στις ε, ε, αξιολογήσεις και διαβεβαιώσεις που δίνονται στους ετήσιους ελέγχους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικούς ελέγχους, ε, καθώς και την γενική έκθεση του εσωτερικού ελεγκτή. Είναι σημαντικός ο ρόλος ε, συνεργασίας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη όπως προβλέπει η συνθήκη, προκειμένου τα κοινοτικά κονδύλια να χρησιμοποιούνται με βάση τις αρχές της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί φυσικά να πραγματοποιεί έλεγχο για το κάθε ευρώ από τα δισεκατομμύρια που καταβάλλονται κάθε χρόνο από το κοινοτικό προπολογισμό. Θα πρέπει να, να στηριχθεί στι διαβεβαιώσει που δίνονται από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση του ισχύοντο μηχανισμού διαβεβαίωση μέσω τη εισαγωγή μιας ετήσιας δήλωσης ε, αξιοπιστίας. Δεν είμαστε κατά της ε, εισαγωγής και μιας πολιτικής δήλωσης για τη διαχείριση των κυρωτικών κονδυλίων, όπως προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Από τις πρόσφατες εμπειρίες που είχαμε ως προς το λογιστικό έλεγχο, τις αιτήσεις εκθέσεις, τις οικειοθελείς ε, αιτήσεις δηλώσεις αξιοπιστίας, Όλα αυτά είναι χρήσιμα στην εσωτερική διαδικασία αξιοπιστία Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα πέρυσι αναλύσαμε τι υπάρχουσες δηλώσει και τι παρουσιάσαμε στα κράτη-μέλη καθώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα σε μια περιεκτική έκθεση με ένα κοινό μοντέλο για το πώ οι εθνικέ δηλώσει αξιοπιστία ε, θα πρέπει να σχηματίζονται και να καταρτίζονται προκειμένου να συμβάλλουν ε, αποτελεσματικά στον, στην αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δυστυχώ δεν έχουν ακολουθηθεί από όλα τα κρατημέλη τα μοντέλα για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστία, αλλά σε τέτοιου είδου έγγραφα πολλέ χώρες δεν εφαρμόζουν το κοινό μοντέλο που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και προτείναμε τη συμπερίληψη μιας διάταξης στον, χρηματο... στον δημοσιονομικό κανονισμό, υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να υποβάλουν κάθε χρόνο και μια διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας. Πρόκειται για ένα μοντέλο που λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί και στα κράτη-μέλη από τις εθνικές διοικήσεις που είναι αρμόδιε για το θέμα αυτό. Όπως είπα παρελειμμένως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί να ενθαρρύνει σε μεταγενέστερη φάση τα κράτη-μέλη για να ε, στηρίξουν πολιτικά τις αιτήσιες ε, ε, δηλώσεις, διαχειριστικές δηλώσεις αξιοπιστίας και στηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο προκειμένου στο δημοσιονομικό κανονισμό να συμπεριληφθεί και μια υποχρεωτική διάταξη για τις εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας που θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επαφείται μόνο στις δηλώσεις των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίσει σωστή διαχείριση και εφαρμογή και αξιοποίηση των κυρωτικών κονδυλίων. Να βάλουμε και από μόνοι μα κάποια μέτρα προκειμένου να ενισχύσουμε την πάταξη τη φοροδιαφυγή. Θα σα αναφέρω τρία τέτοια μέτρα. Καταρχήν, μεταρρύθμιση της νομική βάσης της ΟΛΑΦ. Αναμένεται η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη Ένωση με διατάξει του ποινικού δικαίου και την θέσπιση ενό Ευρωπαϊκού Γραφείου Εισαγγελία. Και μάλιστα οι διαπραγματεύσει για τη μεταρρύθμιση τη ΟΛΑΦ ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και υπάρχουν ε, εύλογε ελπίδε για τη διεκπαιρέωση αυτή τη μεταρρύθμιση στη διάρκεια τη Δανική Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτριά σα, την κυρία Γκρέσλε, που απουσιάζει αυτή τη στιγμή, αλλά εργάζεται πολύ άοκνα και δραστήρια για το θέμα αυτό και ευελπιστώ ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε στι συμβαστικέ λύσει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006. Μάλιστα, ένα από τα βασικά μελήματα του Συμβουλίου είναι να μην ενισχυθεί το γραφειοκρατικό άκθος της ΟΛΑΦ που θα παρεμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία της. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω την υποστήριξή σας και την ελαστικότητα που είναι απαραίτητη για να βρεθεί συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα της μεταρρύθμισης της ΟΛΑΦ. Μάλιστα, για να γίνει πιο αποτελεσματικό το έργο της ΟΛΑΦ, χρειάζεται, όχι, χρειάζεται κάτι περισσότερο από μια απλή αλλαγή της νομικής της βάσης. Χρειαζόμαστε ένα πιο συνεκτικό πακέτο ε, μέτρων, ιδιαίτερα για το ποινικό δίκαιο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ε, και μάλιστα να είναι η προάσπιση αυτή εφάμιλη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην μπορούν δηλαδή ε, να επιλέγουν οι αδικοπρακτούντες μια δικαιοδοσία που θα έχει το χαμηλότερο βαθμό νομικής προστασίας ένα forum shopping. Γι' αυτό και πριν τι θερινέ διακοπέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει μια νέα πρόταση οδηγία για την εναρμόνιση του, του ορισμού των ποινικών αδικημάτων που παραβλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και την εφαρμόσιμη περίοδο περιορισμού. Επίσης, θα θεσπίζουμε ελάχιστες κυρώσεις που θα επιβάλλονται από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση διάπραξης τέτοιων αδικημάτων. Και μάλιστα η οδηγία αυτή θα αντικαταστήσει τους αντίστοιχους, ε, τα αντίστοιχα μέτρα στο, στη Σύμβαση του 1995 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, που προβλέπει ένα πολύ ασθενές επίπεδο εναρμόνισης για να είναι αποτελεσματικό. Η νέα όμως οδηγία θα ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της ε, ενίσχυσης της προστασίας των χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και στο μέλλον. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο του πλαισίου αυτού θα είναι μια νέα νομοθετική πρόταση που θα υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 και θα αφορά την εναρμόνιση των δικονομικών μέτρων. Η πρόταση αυτή στόχο έχει αρχικά την εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν τη χρήση, την συγκέντρωση και χρήση ε, τεκμηρίων και αποδείξεων στις διάφορες διαδικασίες στα κράτη-μέλη και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ε, αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και της ΟΛΑΦ. Και οι δύο οδηγίες ε, θα χαράξουν το δρόμο για μια βελτίωση της προάσπισης των ε, χρηματοοικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και την ανάθεση του σε ένα ειδικό πανευρωπαϊκό εισαγγελικό γραφείο. Μάλιστα, θα υποβάλουμε σχετική πρόταση το 2013 για μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή και θα προβούμε σε μια ε, μελέτη, διεξοδική μελέτη επιπτώσεων, εργασίες τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση αφορά το άρθρο 318 της Ένωσης και υπευλήθη το Φεβρουάριο του 2012, λίγο αργότερα από την αρχικά προβλεπόμενη δηλαδή ημερομηνία. Από φέτο και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να υποβάλει τι εκθέσει αξιολόγηση τη μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου του κάθε χρόνου έχουμε λάβει υπόψη τις αντιδράσεις και τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου μετά την πρώτη έκθεση αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, η φετινή μας έκθεση θα υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση και θα καλύπτει ένα ευρύ, το ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτούνται από τον κοινωτικό προϋπολογισμό και θα περιλαμβάνει και πληροφορίες απόδοσης που θα προκύπτουν από τις αξιολογήσεις και από άλλες αντίστοιχε εκθέσεις. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, ε, το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ένα παράδειγμα απεικοδομητικού και καρποφόρου διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Εκτιμώ ιδιαίτερο την ε, ευκαιρία αυτή που μου δίνεται για ανταλλαγή απόψεων για να ακούσω και τι δικέ σα προτεραιότητε για το 2013 και μάλιστα σε πρόωρο στάδιο. Προσβλέπω λοιπόν με αδειμονία στη συζήτηση και στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς κύριε Επίτροπε που ε, μας διαθέσατε το χρόνο για τις συζητήσεις μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχω αρκετούς συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις, όμως θα ήθελα να εκμεταλλευτώ το προνόμιο που έχω σαν Πρόεδρος για να επανέλθω σε ένα σημείο που μόλις αναφέρατε, τον Ευρω... την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Ξέρουμε ότι το προωθεί η Βιβιάνε Ρέντινγκ, η συνάδελφός σας, και το συζητήσαμε εδώ και στην Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών. Όμως αυτό το θέμα πάντα ήταν ένα θέμα σημαντικό για την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, δηλαδή προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ερώτηση. Έχετε ακριβές χρονοδιάγραμμα που θα μπορούσατε να μας κοινοποιήσετε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ποια είναι η εντύπωσή σας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να συνεργαστεί με την αρμόδια επιτροπή επί του θέματος αυτού. Θα μετακινήσω το βάρος προς τα δικαστικά θέματα, τα νομικά θέματα, ή σαν επίτροπος θεωρείται ότι αφορά περισσότερο ε, την, τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό σημαντικό χαρτοφυλάκιο και όπως είπα και στην εισαγωγή μου, οι υπηρεσίες μας ξεκίνησαν αξιολόγηση συνεπιών, αναλύοντας διάφορες επιλογές, διάφορες δυνατότητες, οι οποίες θα αξιολογηθούν με αντικειμενικά κριτήρια. Και βάσει της αξιολογήσεως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει την προσέγγισή της. Θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια μορφή θα έπρεπε να έχει στο μέλλον. Αυτή η υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελία, είναι αρκετά φιλόδοξο σχέδιο. Η ιδέα είναι να αποβληθεί τον Μάιο του 2013 το σχέδιο, ήδη. Καταρχάς βέβαια πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση αντιχτύπου και πιστεύω ότι θα διεξαχθούν εις βάθος συζητήσει επί συγκεκριμένων στοιχείων της προτάσεως. Θα συζητηθεί και εδώ, στο Κοινοβούλιο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάν Μούλτερ ήταν ο πρώτος που ήθελε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δράτω με τις ευκαιρίες να συγχαρώ τον Επίτροπον για αυτά που είπε στην ε, Ολομέλεια για τις ετήσιες συνόψεις. Η δήλωσή του ήταν άκρος ευπρόσδεκτη από την Επιτροπή μας και από το Κοινοβούλιο Γέννη. Είναι ο πρώτος επίτροπος, πιστεύω, στα έξι χρόνια που κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση για την εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας του 2006. Νομίζω ότι είναι ντροπή που το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν έτοιμοι νωρίτερα να κάνουν αυτά που κατά την άποψη του Κοινοβουλίου είχαν συμφωνηθεί και ήταν ξεκάθαρο. Αν γίνει συμφωνία μεταξύ τριών μερών για κάποια σύνοψη που θα πρέπει να συντάσσεται, τότε κατά την άποψή μου εξυπακούεται ότι αυτή η σύνοψη διατίθεται και για τα τρία μέρη. Η μη η απόφαση ήταν διαφορετική. Επί έξι χρόνια και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερναν να προβάλλουν διάφορα επιχειρήματα προς το Κοινοβούλιο και να τον μπερδεύουν. Αυτό ήταν θαύμα θα έλεγα, αλλά χαίρομαι που έθεσε τέρμα στην κατάσταση ο Επίτροπος. Τι θέλουμε, θέλουμε να έχουμε τις αιτήσεις συνοπτικές σε αυτές εκθέσεις. Θα θέλαμε να έχουμε τα σχόλια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποιο είναι το θέμα, ότι δεν υπάρχει αρκετός δημοκρατικός έλεγχος όσον αφορά τα 80% των χρημάτων που δαπανούν τα κράτη-μέλη. Εμείς, σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα κράτη-μέλη. Αυτό θα πρέπει να αναλυφθεί από τα Εθνικά Κοινοβούλια, τα οποία δεν το κάνουν. Τι ο τρόπος όμως μπορούμε να καλύψουμε το δημοκρατικό κενό. Ο καλύτερος τρόπος είναι οι εθνικές δηλώσεις. Τι ο τρόπος αναλαμβάνεται πολιτική ευθύνη και τα κράτη-μέλη θα μας δείχνουν ποιος είναι πολιτικά υπεύθυνο, διότι θα ετοιμάζει δήλωση. Αν κάποιος ετοιμάσει δήλωση που είναι αναλυθής, θα ξέρει αυτός που το κάνει ότι δεν κάνει καλό για το πολιτικό του μέλλον. Και γι' αυτό η, η εθνική δήλωση θα είναι μια πολιτική δήλωση επίσης. Και θα καλύπτει το δημοκρατικό κενό. Για να το πετύχουμε αυτό, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δίνει και κίνητρα και κυρώσεις. Δηλαδή τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία ε, δίνουν μια εθνική δήλωση, αν η εθνική δήλωση αυτή είναι ορθή και το διαπιστώσει αυτό το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί αυτή την περιπτώση, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να ελέγξει περισσότερο τα άλλα κράτη-μέλη τα οποία δεν χορηγούν αυτή την εθνική δήλωση. Θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική ξύλου και καρότου κινήτρων και ποινών. Αυτή είναι η ουσία των όσων αντικατοπτρίζονται στα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης όμως και στην πρόσφατη ψηφοφορία για το δημοσιονομικό κανονισμό που διαπραγματευόμαστε, το είδαμε. Ε, παρατηρήσαμε από ότι κάποια κράτη-μέλη ήθελαν να επαναχωρήσουν και από αυτά που συμφωνήθηκαν στη Διοργανική Συμφωνία του 2006. Και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν λοιπόν προς τα κράτη-μέλη ότι δεν θα υπαναχωρήσουμε σε κάτι που ήδη έχει συμφωνηθεί προεξαετίας. Αυτός είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πετύχει θετική δήλωση ε, αξιοπιστίας. Θα έλεγα λοιπόν, απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγχαρητήρια και συνεχίστε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, ευχαριστώ, συνάδελφα Γιάνν Μούλτερ. Άλλος ένας συνάδελφος και μετά θα δοθούν οι απαντήσεις. Ο Ζαν Πιεροντή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτό το διάλογο που έχετε με την Επιτροπή μας. Μιλάμε για προγράμματα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2013. Το 2013 είναι τελευταία πλήρης χρονιά της παρούσης θητείας, διότι η εντολή της θητείας τελειώνει το 2014, όπως και δική μας και θα μπούμε στη χρονιά των διαπραγματεύσεων των δημοσιονομικών προπτικών και διαρωτώ με μήπως θα ήταν η καλή στιγμή να κάνουμε μία εξέταση γενική θα έλεγα να δούμε τι δουλεύει, τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά. Διότι έχουμε πολλές τέτοιες συναλλαγές, πολλές γενικές συζητήσεις ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία είχε πει ότι σας εγγυώμαι ότι θα υπάρξει θετική δήλωση αξιοπιστίας. Ο συνάδελφος αναφέρθηκε στη θετική δήλωση αξιοπιστίας. Εγώ δεν ξέρω τι είναι η θετική δήλωση αξιοπιστίας. Διαβάζω τα συμπεράσματα της εκθέσεως, τα πορίσματα της εκθέσεως του ελεκτικού συνεδρίου δεν ξέρω αν είναι αρνητική δήλωση εξοπιστία, αν είναι αποχή από γνωμοδότηση, δεν ξέρω αν θετική δήλωση εξοπιστία, δεν ξέρω πλέον ποιο είναι ο στόχο μα. Διερωτώ με μήπως ήρθε η στιγμή να τα θέσουμε όλα επιτάπητος μαζί με τα κράτη-μέλη, με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε τα τελευταία 15 χρόνια και να πούμε τι κάνουμε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, μήπως θα έπρεπε να δούμε αν μπορεί να υπάρχει καλύτερη συνεργασία με εθνικούς φορείς, εθνική εξουσία, εθνική διοίκηση, τοπική ε, ε διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ευρωπαϊκή διοίκηση για να χειριστούμε την Ήπειρο. Περνάμε μια πολύ δύσκολη ε, κρίση και όλοι φυλάζουν ε, τα, τα δικά τους προνόμια, τοπική αυτοδιοίκηση, εθνική διοίκηση, ευρωπαϊκή και ο καθένας διαφυλάσσει τα συμφέροντά του και δεν υπάρχει συνολική ε, συνοχή. Αναφερθήκατε σε αυτή την ετήσια δήλωση για τη διαχείριση. Εγώ δεν πίστεψα ποτέ, αντίθετα από τους συναδέλφους σε αυτήν την Επιτροπή, ότι θα είχαμε πολιτικές δηλώσεις αρχηγών κρατών ε, που εξάλλου δεν είναι ο ρόλος τους να κάνουν δηλώσεις όσον αφορά τους ελέγχους. Εκεί είναι για να ασκούν την πολιτική και εμείς είμαστε εκεί για να ελέγχουμε, να ελέγχουμε. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη δήλωση διαχείριση. Σα κάνω μια πρόταση κύριε Επίτροπε αν μπορείτε να πείσετε αυτού που είναι γύρω σα, να συνοδεύετε αυτή η δήλωση της διαχείρισης, διαχειριστική δήλωση, από μια βεβαίωση ελέγχου των Εθνικών Ελεκτικών Συνεδρίων που θα δήλωναν ότι αυτή η ετήσια ε, διαχειριστική δήλωση είναι μια λογική διαβεβαίωση ή ότι στην κοινή διαχείριση τα έκαναν σωστά, σεβάστηκαν τους κανόνες τα κράτη και ότι αυτές δηλώσεις γίνονται ειλικρινώς και εμείς θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητη άποψη που θα έχει αξία έλεγχου, διότι αυτές οι εθνικές δηλώσεις που ζητούμε έχουν μια αξία στον αφορά τους ελέγχους, τη, διαδικασία, Α, και, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η προσέγγιση σωστή. Θέλω πριν το τέλος της θητείας μας να δούμε, να εκμεταλλευτούμε τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες μας, να δούμε αν θα συνεχίσουμε με τα συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε τώρα. Εγώ θα πρότεινα Μήπως ήρθε στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει χρηματοστατική διοίκηση. Για την ώρα έχουμε κοινή διαχείριση. Γιατί, διότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να έχουμε τη δική μας χρηματοστατική διαχείριση. Γιατί εμείς να μην έχουμε με τέτοια διοίκηση αντί να αναθέτουμε αυτή την κοινή διαχείριση στα κράτη-μέλη. Θα έκλεινα λέγοντας ότι το θέμα του φθινοπόρου ομιλία για την κατάσταση που κρατεί στην Ένωση, που θα, ομιλία που θα δώσει ο πρόεδρος Μπαρόσο, θα εισακουστεί όλος ιδιαίτερος, θα είναι δεδομένη κρίσιμη στιγμή που αφορά την Ένωση. Λοιπόν, όταν ε, ξεχνιάζουμε τι είπε, αναφέρθηκε στον έλεγχο πολύ στην προηγούμενη, αναφέρθηκε πολύ στην προηγούμενη θητεία. Ελπίζω ότι χάρη στη δουλειά που κάνετε και στις παρατηρήσεις που σας κάνουν οι βουλευτές επιτροπές ελπίζω ότι ο πρόεδρος Μπαρόσο θα έχει μία παράγραφο που θα αναφέρεται στους ελέγχους ε, θα αναφέρεται στο όραμα όσον αφορά τη λειτουργία την οικονομική, τη χρηματοστοτική των δημοσιονομικών τι γίνεται με τις δαπάνες, τα κράτη-μέλη ποιο συντονισμό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει συμπληρωματικότητα και όχι αντίθεση μεταξύ ευρωπαϊκού επίπεδου και εθνικού επίπεδου ε, ζητώ συγγνώμη που του χρόνου το θέμα τη Ελληνική Ένωση. όλες οι εκθέσει του ελεκτικού συνεδρίου και οι πληροφορίε που μα δίδονται δείχνει ότι λειτουργεί άσχημα η Τελωνιακή Ένωση. Αν έχουμε μια αρμοδιότητα, είναι πράγμα Τελωνιακή Ένωση όμω. Στι συνθήκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαν αρμοδιότητα αποκλειστική την Τελωνιακή Ένωση. Μήπω δεν ήρθε η στιγμή να μελετήσουμε ε, αν μια πρόταση που έγινε πριν 4-5 χρόνια ε, να έχουμε Ευρωπαίου υπαλλήλου που ασχολούνται με την Τελωνιακή Ένωση. Δηλαδή πώ λειτουργούν τα τελωνία. Να ελέγχονται από την Ένωση ιεραρχικά και όχι από τα κρατη διότι βλέπουμε ότι όλες οι δυσλειτουργίες που έχουμε όσον αφορά την Ένωση οφείλονται στο ότι αναθέτουμε αυτά τα καθήκοντα στα κράτη-μέλη. Είτε αφορά το Σέγγεν για κάποια σύνορα, τελωνιακή ένωση, για τη χρηματοδοτική λειτουργία. Μήπω επί κάποιων λειτουργιών, τουλάχιστον αποκλειστικών, δεν θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μελετήσουμε το ενδεχόμενο να υπάρχουν υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διαχειρίζονται την πολιτική λειτουργία, την απο, τις αποκλειστικές αυτές λειτουργίες που έχουμε και καθήκοντα ξεκινώντας την Τελωνιακή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, Κύριε Οντή, πραγματικά ήταν πολύ σημαντικές αυτές οι ερωτήσεις όπως και αυτές του κύριου Μιλντερ και θεωρώ πως ε, έχουμε αρκετά θέματα για να απαντήσει ο κύριος Επίτροπος. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είδα πως ο Γιάνν Μιλντερ άργησε λίγο να μπει στην αίθουσα. Στην αρχή αναφέρθηκα στις ε, δηλώσεις και σε αιτήσιες συνόψεις ε, των κρατών μελών και τις συνόψεις αυτές ε, συμπεριλαμβάνουν και σχόλια της Κομισιόν επί τη βάση των ε, αιτήσεων ε, εκθέσεων δραστηριότητας της ε, Γενικής Διεύθυνσης, αλλά σκοπεύουμε βεβαίω να κάνουμε πιο συνολική αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών συνόψεων και στα μέλη της Επιτροπής κατόπιν και οι δύο αναφέρατε το θέμα των δηλώσεων είτε διαχειριστικών είτε εθνικών και νομίζω πως αυτό το είναι σημαντικό τώρα είναι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να βρούμε τη λύση και να συμπεριληφθούν αυτές οι απαιτήσει στον δημοσιονομικό κανονισμό γιατί χωρίς τον κανονισμό βεβαίως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε απαιτήσει από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώς οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται για το δημοσιονομικό κανονισμό είναι πολύ κρίσιμες και για να αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα του ελέγχου αυτό το οποίο προτείνουμε είναι αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Οντί. Προτείνουμε δηλαδή διαχειριστικές δηλώσεις ε, αξιοπιστίας μαζί με ελεγκτικές δηλώσεις, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε να βάλουμε στον κανονισμό την απέτηση οι ελεγκτικές αυτές δηλώσεις ε, που πρέπει να, γίνουν, ναι, να πρέπει να γίνουν από τα ανώτατα ελεγκτικά όργανα γιατί είναι και ζήτημα ε, κυριαρχίας και ανεξαρτησίας των οργάνων αυτών αλλά εγώ εκμεταλλεύομαι κάθε ευκαιρία για να συναντηθώ με επικεφαλής των ανώτατων ελεγκτικών οργάνων και τους ε, ζητώ αυτοί να αναλάβουν ευθύνη και να ε, ελέγξουν τις ε, ετήσιες δηλώσεις διαχείρισης. Αυτό σχεδιάζουμε τώρα, αλλά βεβαίως το πιο σημαντικό ζήτημα από πολιτική σκοπιά είναι να υιοθετηθούν αυτές οι διατάξεις στον δημοσιονομικό κανονισμό. Όσον αφορά τώρα μαστίγια και καρότα που αναφέρατε σε σχέση με αυτούς που εθελοντικά κάνουν εθνικές πολιτικές δηλώσεις είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να εξετάσουμε βεβαίως αυτή τη στιγμή ελάχιστα είναι τα κράτη-μέλη, είναι τέσσερα αυτά τα οποία κάνουν εθνικές δηλώσεις και μόνο ένα από αυτά κάνει μια δήλωση η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσει της ε, Κομισιόν. Αν το κάνουν και άλλα ε, κράτη-μέλη, να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να τους ε, ενθαρρύνουμε στο πλαίσιο αυτό του έλεγχου. Κατόπιν το ζήτημα της ε, Τελωνιακής Ένωσης. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αξιολογήσουμε την ε, Τελωνιακή Ένωση και είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται ούτως ή άλλως οι υπηρεσίες μας ε, προετοιμάζουν ε, την ε, λεγόμενη ανακοίνωση που λέγεται η κατάσταση της Τελωνιακής Ένωσης. Πρόκειται για μια αξιολόγηση της Τελωνιακής Ένωσης που προβλέπεται να γίνει στο τέλος του έτους και στόχος είναι να δούμε την κατάσταση στην Τελωνιακή Ένωση και ελπίζω να κάνουμε και κάποιες συστάσεις για το πώς θα προχωρήσουμε. Οπότε δεν θέλω τώρα να προκαταλάβω κάποια απόφαση που θα λάβουμε γιατί οι υπηρεσίες μας αυτή τη στιγμή αξιολογούν την κατάσταση. Και όσον αφορά την ομιλία του Προέδρου της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης. Ε, δεν μπορώ να σας υποσχεθώ συγκεκριμένη αναφορά στην ομιλία του κυρίου Μπαρόζο αυτή τη στιγμή, αλλά πρέπει να πω πως ε, παραδείγματος χάρη η συνθετική αυτή η έκθεση αποτέλεσε μέρος ε, προφορικής συζήτησης ε, εντός της Επιτροπής και ε, θα γίνει νομίζω ούτως ή άλλως την Τετάρτη θα επαναληφθεί μια τέτοια συζήτηση. Οπότε ο έλεγχος είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το δούμε και πολιτικά και να δούμε τι μορφή θα έχει βεβαίως η ε, ομιλία του κυρίου Μπαρόζο. Αυτό είναι δική του απόφαση. Οπότε, νομίζω πως κάλυψα Α, ναι. Με συγχωρείτε. Για το θέμα που ορίσατε ως επιστροφή στις ρίζες και να ξαναδούμε τους κανόνες. Νομίζω πως τώρα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία γιατί συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και οπωσδήποτε οι κανόνες οι οποίοι προτείνονται για διάφορα προγράμματα θα μπορούν να αξιολογηθούν λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας που έχουμε ήδη εδώ και πολλά χρόνια και η θεωρεί πως μάθαμε πολλά την εμπειρία μας και οι νέοι κανόνες που προτείνουμε ακριβώς αντιμετωπίζουν όλα σχεδόν τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην ε, διαδικασία της απαλλαγής από τους ελέγχους του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά βεβαίως η συζήτηση με το Συμβούλιο μπορεί να μας δώσει κάποια περιττέρω στοιχεία και έχουμε ένα κοινό στόχο δηλαδή οι κανόνες ε, για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να είναι απλοί, αποτελεσματικοί και να δίνουν τη δυνατότητα πρόληψης των ε, λαθών και της απάτης. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δύο συνάδελφοι ακόμα, η Ινές Αγιάλα Σέντερ και μετά Γιένς Γκάιερ. Ινές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Σεμέτα και στερνίζομαι πλήρως και τα, σχόλια του Προέδρου καθώς και τα σχόλια του κυρίου Μίλντερ σε ό,τι αφορά τις α, συνόψεις, συνοπτικές εκθέσεις για τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την απαλλαγή του Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σε διέξοδο ως προς αυτή την απαλλαγή και παρά τις αγαθές προθέσεις και την καλή θέληση της Δανικής Προεδρίας, δυστυχώς δεν σημειώσαμε καθόλου πρόοδο και όλο και περισσότερο ακούγεται η άποψη ότι μία πιθανή διέξοδος με την οποία δεν συμφωνώ αλλά φαίνεται ότι γίνεται η κρατούσα άποψη είναι και το συζητά και το Συμβούλιο μία διέξοδος να προέλθει από την ανάκτηση της ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή να αναλάβει την ευθύνη και να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε και η Κομισιόν ως αρμόδια για την απαλλαγή αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπαμε και για τις συνόψεις, ε, να ενημερώνεται εγκαίρως και εκτεταμένα για ένα θέμα για το οποίο και εμείς είμαστε αρμόδιοι, όπως είναι το θέμα της απαλλαγής. Ερωτώ λοιπόν κύριε Σεμέτα. Μας είπατε σήμερα ότι καταφέρατε επιτέλους και βρήκατε και μας επιδώσατε τι συνόψει των κρατών μελών. Θα μπορούσε κάτι αντίστοιχο να γίνει και για την απαλλαγή του Συμβουλίου, να σημειωθεί και εκεί πρόοδος και να διέλθουμε από το αδιέξοδο. Σε ό,τι αφορά τον δημοσιονομικό κανονισμό, γιατί φαίνεται ότι είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα. Πώς μπορούμε ε, να προωθήσουμε πρόοδο στο θέμα της απαλλαγή, χρησιμοποιώντας κατά κάποιο τρόπο το δημοσιονομικό κανονισμό. Προσπαθώντας έτσι να κινητοποιήσουμε το Συμβούλιο. Και κάτι άλλο που υπενηχθήκατε κι εσείς. Φαντάζομαι θα το θίξει και κάποιος συνάδελφος για τους ίδιους πόρους. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγέ. Το νέο ΦΠΑ, το θέμα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Αλλά και ως προς το ζήτημα των δημοσιονομικών προοπτικών. Αρχίζει η προετοιμασία για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Λάβαμε την πρωτόλαιο πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι, μέχρι ότου όμως διεκπαιρεωθεί το θέμα και μέχρι να αρχίσει το 2014. Εσείς ως αρμόδιος επίτροπος έχετε προβλέψει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τις επιστροφές, για την ε, κακή η μη χρήση των, του προπολογισμού από τα κράτη-μέλη, γιατί κάνουν υπερεκτίμηση των αναγκών, δεν εξαντλούν το προπολογισμό και προσπαθούν να, το, να κρατήσουν αυτά τα κονδύλια στα ταμεία τους. Αυτές τις δυσλειτουργίες του προϋπολογισμού πώς θα τις αντιμετωπίσετε. Γιατί υπάρχουν όντως προβλήματα και ίσως με κάποια βελτίωση στον μηχανισμό θα μπορούσαμε από την αρχή να τα εξαλείψουμε. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κυρία Αγέλα. Σέντερ, ο κύριος Γκάιρ. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη γιατί έφυγα στις 5.30 ε, η ώρα. Ο επικεφαλής συνοβουλευτικής μας ομάδας ε, στην ε, Γερμανική Βουλή βρισκόταν εδώ πέρα και είμαι υπεύθυνο για αυτές τις επαφές, οπότε ήταν ανηλυμένη η υποχρέωση. Και ήθελα να αποφύγω αυτό το οποίο συχνά βλέπω εδώ μέσα, να γίνονται ερωτήσεις και μετά να μην βρίσκεται εδώ πέρα ο βουλευτής να ακούσει την απάντηση. Να αναφερθώ τώρα σε αυτό που είπε η Ίνες. Θεωρώ πως έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία στον έλεγχο των δημοσίων ευρωπαϊκών οικονομικών να προχωρήσουμε αν το συνδυάσουμε με τη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο οικονομικό πλαίσιο. Ζούμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη είτε λένε πως θα θέλαμε περισσότερα κονδύλια από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό είτε αυτό το οποίο λένε οι καθαροί εισφορείς, δηλαδή η Γερμανία ας πούμε η χώρα μου όπου λένε καλύτερα λιγότερα, αλλά οπωσδήποτε όχι περισσότερα. Σε μια τέτοια λοιπόν κατάσταση, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο αν ε, κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, τη στιγμή στην οποία συζητάμε ποιες ε, αρμοδιότητες έχουν τα κράτη-μέλη για την απάτη ΦΠΑ, για τους τελωνιακούς ελέγχους. Επιτυγχάνουμε δύο πράγματα. Επιτυγχάνουμε αποτελεσματικό έλεγχο των ε, ίδιων ε, πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ε, τελικά θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε περισσότερους ίδιους πόρους από αυτές τις πηγές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσως εδώ πέρα η Κομισιόν μπορεί να κάνει κάποιες εκτιμήσεις σε ποιο βαθμό ήδη αυτοί οι πόροι μπορούν να επεκταθούν δηλαδή τι περισσότερο θα είχαμε με περισσότερους ελέγχους και από την άλλη τα κράτη-μέλη λένε κοιτάξτε να δείτε άμα θέλετε αν έχουμε αποτελεσματικούς ε, ελέγχους ε, θα έχουμε νομίζω και περισσότερα έσοδα. Οπότε νομίζω πως με το ζήτημα της αποτελεσματικότητας ε, θα έχουμε ένα μοχλό αν θέλετε για αυτή την συζήτηση. Και θα χαιρόμουν κύριε Επιτροπέ αν μπορέσουμε να συνεργαστούμε από κοινού αποτελεσματικά για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και να δείξουμε πως ε, τα κράτη-μέλη πράγματι ελέγχουν ε, και θέλουν να ενισχύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πάνω στην ώρα ήρθε και η κυρία Γκρέσλε. Έχετε το λόγο. Με συγχωρείτε που δεν παρακολούθησα τη συζήτηση, αλλά ε, ο πρόεδρος ε, της κοινοβουλευτικής ομάδας μας ε, στην Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή βρίσκεται και εμάς εδώ πέρα και των Σοσιαλδημοκρατών και των, και των Χριστιανοδημοκρατών και έχω να σας πω κάτι το σημαντικό που αφορά τον ε, μελλοντικό επίτροπο από την Κροατία. Κύριε Σέμετα, εσείς έχετε ένα τεράστιο χαρτοφυλάκιο και όλοι υποθέτουν πως θα μοιραστεί. Να σας πω πως, εάν κάποιος ε, είχε την ιδέα να δώσει το χαρτοφυλάκιο της απαλλαγής στον ε, νέο επίτροπο, εγώ θα ήμουν κατά η ομάδα μου βεβαίως θα ήταν κατά. Σας ε, ευχαριστώ για τη συμμετοχή σε συζήτηση. Τώρα ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω διότι μου ετέθησαν πολλές ερωτήσεις όσον αφορά τους ίδιους πόρους. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να προωθεί αυτό το καθεστώς των ιδίων πόρων και για το ΦΠΑ και για το φόρο χρηματοσυντικών συναλλαγών. Θα δεξαχθεί η πολιτική συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ όσον αφορά το φόρο χρηματοστικών συναλλαγών στις 22 Ιουνίου όπου θα δούμε ποια θα είναι τα επακόλουθα βήματα. επεξεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη δυνατότητα συμβιβασμού, αλλά δεν τα καταφέραμε ακόμα. Έτσι έχουν τα πράγματα όσον αφορά το φόρο επιχειρηματικών συναλλαγών, όσον αφορά το ΦΠΑ ιδίου πόρους, είναι πιο εύκολη η κατάσταση. Πολλά κράτη-μέλη υποστηρίζουν τις ιδέες που παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη αλλά για τους ιδίους πόρους χρειάζεται η ομοφωνία και επικύρωση από τα κράτη-μέλη. Δεν είναι εύκολη η διαδικασία. Εξακολουθούμε όμως να το προωθούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι οι ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πραγματικοί ίδιοι πόροι, θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν τις διατάξεις της συνθήκης Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να χρηματοδοτείται από τους ιδίους πόρους, ενώ μέχρι τώρα είχαμε 75% συνεισφορές από τα κράτη-μέλη. Τώρα, όσον αφορά απάτες και αποφυγή τους, έχουν ύψιστη προτεραιότητα αυτά για φέτος. Ετοιμάζουμε την έκθεση που ευβοληθεί στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό του Ιουνίου. Εκεί θα παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις για μέτρα αντιμετωπίσεως των απατών και τρόπους αποφυγής των απατών. Προτάσεις που σχετίζονται με απάτη στον τομέα του ΦΠΑ Αυτό άπτεται και των τελωνιακών σε κάποιο βαθμό. Θέματα λαθρεμπορίου είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Προτιθέμεθα να παρουσιάσουμε σχετικούς ιδέες. Αργότερα, φέτος, θα υποβάλουμε μια ανακοίνωση. Η ανακοίνωση θα παρουσιάζει πλήρη κατάλογο μέσων τα οποία θα επιτρέψουν καλύτερη καταπολέμηση των απατών στον τομέα του, των φόρων και την φοροδιαφυγή. Αυτά είναι στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, είμαι υπεύθυνο για τα θέματα των φόρων και αυτές οι συνδέσεις που αφορούν περισσότερο αυτά τα θέματα, αλλά συνδέονται και με τα έσοδα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Επισήμως παρουσίασα τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαλλαγή του Συμβουλίου και επί χάρτου παρουσίασα την τοποθέτησή μου. Διεξήχθη πολύ καλή συζήτηση μαζί σας. Συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια κάποια πρόοδο. Καλύτερη λύση θα ήταν και οι δύο κλάδοι του προπολογισμού, οι δύο αρχές του προπολογισμού να συμβιβαστούν. Γιατί είναι ευαίσθητο το θέμα αυτό. Η συνθήκη αναφέρει ξεκάθαρα ποιο είναι ο ρόλος του Κοινοβουλίου και ότι το Κοινοβούλιο είναι η αρχή αρμόδια για την απαλλαγή για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κανονικά το θεσμικό όργανο που παρέχει συμβουλές επί διαφόρων θεμάτων, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ήταν δύσκολο να δώσω περισσότερες συμβουλές από αυτές που ήδη έδωσα κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. Ο κύριος Γκάιερ έχει απόλυτο δίκιο. Αν μπορούσαμε να έχουμε, να έχουμε καλύτερη συλλογή ε, των εσόδων, θα είχαμε μείωση της συνεισφοράς των ε, κρατών μελών. Θα ήταν ένα καρότο δηλαδή προς τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες που καταβάλουν για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Να πω επίσης ότι θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπάρχοντα μέσα που προβλέπει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντάσσουμε εκθέσεις για το τι γίνεται με τη συλλογή του ΦΠΑ στα διάφορα κράτη-μέλη και στην επόμενη έκθεση πρόθεσή μας είναι να κάνουμε μια βαθμολόγηση των κρατών μελών να δείξουμε ποια είναι η αποδοτικότητά τους όσον αφορά τη συλλογή του ΦΠΑ αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει τη δραστηριοποίηση της προσπάθειας καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Είναι σαφές ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αυτό το τομέα του ΦΠΑ. Υπάρχουν ε, μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων για τη συλλογή του ΦΠΑ, για την ίσπραξη του ΦΠΑ. Μετά, το θέμα του Κροάτη Επιτρόπου. Δεν θέλω να σχολιάσω. Αυτό είναι ευθύνη του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείνος μοιράζει τα καθήκοντα, εκείνος αναθέτει τα καθήκοντα στους νεοδιοριστέντες επιτρόπους. Δεν θα ήθελα να κάνω συγκεκριμένες προτάσεις στον Πρόεδρο. Ο πρόεδρος αποφασίζει το πώς θα χειριστεί το θέμα. Εν συντομία, αυτές τις απαντήσεις ήθελα να δώσω στις τελευταίες αυτές ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, είμαι έτοιμος να απαντήσω και αυτές. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε εξ ονόματος ε, της ε, Επιτροπής μας για το ότι απαντήσατε στις ερωτήσεις αυτές. Εκτιμούμε το ότι υπάρχει τόσο καλή συνεργασία και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο Γιάνν Μούλτερ. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό το ότι πήρατε τις αιτήσει ε, συνόψεις και τις παρουσιάσατε σήμερα. Είναι απαράδεκτο το ότι χρειάστηκαν 6 χρόνια, αλλά είναι θετικό το ότι τα καταφέρατε. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με την κυρία Γκρέσλε και ίσως μπορείτε να μεταβάσετε στους άλλους ε, επιτρόπους πως ε, ο πρόεδρος Μπαρόζο και η υπόλοιπη επιτροπή καλά θα κάνει να λάβει υπόψη τη γνώμη της επιτροπής μας. όσον αφορά το ποιο ο Επίτροπος θα είναι αρμόδιο για την απαλλαγή και να λάβετε ίσω και υπόψη την άποψή μα για το ποιο θα πρέπει να είναι αυτό ο επίτροπο. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συζήτηση, για το ότι απαντήσατε ε, στις ερωτήσεις μας και για το ότι είστε ο επίτροπο ο αρμόδιος ε, για το θέμα αυτό και σε συνεχή επαφή ε, με την Επιτροπή μας.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 από τη συνάδελφοι, προχώρησε λίγο παραπέρα η διαδικασία. Καθυστερήσαμε και με την ακρόαση και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση του Τόμας Ντόιτς για την ενίσχυση της κανότητας Κροατίας όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις μετά την ένταξη. Οπότε Καλωσορίζω επίσης ε, και τον κύριο Φαζάκας, ε, μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Χαίρομαι που είστε εδώ. Δίνω το λόγο στον ε, εισηγητή μας λοιπόν πρώτα, τον κύριο Ντόιτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ τον εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, τον κύριο Φάζακας. Και να πω ότι το σχέδιο έκθεσης μας καλύπτει την ειδική έκθεση 14 του 2011 του Ελεκτικού Συνεδρίου και αυτή η ειδική έκθεση έχει τίτλο «Έχει η, ε, η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βοηθήσει την Κροατία να διαχειριστεί τα με τα ενταξιακά κονδύλια. Εν είδη εισαγωγής, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι μιλούμε εδώ για ένα πολύ ευρυθμό σύστημα. Το σύστημα και ο μηχανισμός που διέπει την ένταξη μιας χώρας καθ' όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας είναι πολύ αποτελεσματικό. Είναι μια πολύ καλά ε, λειτουργούσα και εύρυθμη διαδικασία από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέχρι την ε, επίσημη προσχώρηση μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μάλιστα εκπροσωπώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια χώρα που πριν από 10 χρόνια πέρασε από την ίδια αυτή ε, ενταξιακή διαδικασία και γνωρίζω εκ πείρας ότι δύο είναι τα τεινά που θα πρέπει να αποφύγουμε στη διαδικασία αυτή. Αν έχουμε κράτη-μέλη που διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις σε διαφορετικό χρονικό διάστημα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και σταθμά για να αξιολογούμε τις επιδόσεις ε, των χωρών αυτών. Θα πρέπει τα ίδια κριτήρια να εφαρμόζονται για όλους. Και ανέκαθεν προσπαθούσαμε να αξιολογήσουμε τις επιδόσεις και την οριμότητα μιας επίδοξης ε, ε, για ένταξη χώρας, μιας υποψήφιας για ένταξη χώρας και οι προϋποθέσεις της προσχώρησης κατοχυρώνονται σε νομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν πολύ πριν από τη συγκεκριμένη υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και εδώ στην περίπτωση της Κροατίας και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι ακόμη και αν η ενταξιακή συμφωνία υπεγράφει μόλις πέρυσι το Δεκέμβριο, Εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο μία επιτροπή αξιολόγησης και αυτή η επιτροπή αξιολόγηση εξέτασης αξιολογεί τις επιδόσεις μιας χώρας μετά την αποδοχή της, ε, της υποψηφιότητας της χώρας αυτής. Αλλά παραλαμβάνω δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαφορετικά μέτρα και σταθμά για τις ε, διαδοχικές διευρύνσεις. Η τήρηση των κανόνων δεν είναι μόνο προς το συμφέρον τη ενδιαφερόμενη χώρα, είναι και προς το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 2010, το 2004, συγγνώμη, είχαμε ένα σημαντικό γύρο διευρύσεων προς 10 νέες χώρες, κάτι που ενίσχυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν απέβη μόνο προς όφελος των 10 νέων χωρών, αλλά και τη παλιά Ένωση. Το ίδιο ισχύει και για την υποψηφιότητα της Κροατία σήμερα. Θα εξυπηρετήσει όχι μόνο την Κροατία, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έρθω τώρα στις συγκεκριμένες συστάσεις και το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Σε ό,τι αφορά τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει, αυτέ ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία ημέρα τη Ουγγρική Προεδρία, πέρυσι δηλαδή, πέρυσι το Δεκέμβριο συγκεκριμένα, τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε την ενταξιακή συμφωνία με την Κροατία. Και σε λιγότερο από 13 μήνες η Κροατία θα γίνει και επίσημα το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κροατία υποφελήθηκε από πολλά είδη χρηματοοικονομικής συνδρομής τα τελευταία χρόνια και ο λόγος που παρέχουμε αυτή την ε, συνδρομή είναι για να προετοιμάσουμε την υποψήφια χώρα για την ένταξή της. Θέλουμε να βεβαιωθούμε βέβαια ότι η συνδρομή αυτή χρησιμοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξιοποιήθηκε στο έπακρο. Τον έλεγχο αυτό διενήργησε το ελεκτικό συνέδριο και τα απορίσματά του περιλαμβάνονται στην ε, ειδική αυτή έκθεση. Καθ' όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αξιολόγησης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολούθησε την όλη διαδικασία και πρόσφατα δημοσίευσε και την έκθεσή της, την έκθεση παρακολούθησης ε, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και η ειδική έκθεση του Ελεκτικού συνεδρίου για την Κροατία, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η προενταξιακή αυτή διαδικασία εξυπηρέτησε την Κροατία και την και ενίσχυσε την δυνατότητά της και την ικανότητά της να διαχειριστεί και την μετενταξιακή χρηματοδότηση. Και οι δύο εκθέσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεκτικού Συνεδρίου επισημαίνουν διάφορους τομείς που χρήζουν περαιτέρω πρόοδου. Για παράδειγμα αναφέρονται οι εκ των προτέρων έλεγχοι η έλεγχοι εξάντε που θα πρέπει να παραμείνουν ενισχύ και στο μέλλον μετά την προσχώρηση της Κροατίας και επίσης οι κροατικές αρχές θα πρέπει να ενισχύσουν τη δυνατότητα απορρόφησης, ε, την ικανότητα εκταμίευσης ε, των κοινοτικών κονδυλίων και φυσικά να ενισχύσουν την πάταξη της δωροδοκίας και της διαφθοράς. Η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου επισημαίνει ότι οι δικαιούχοι της Συνδρομής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οικονομικής αυτής αρρωγής και οι αρμόδιοι για τη διαχείριση αυτής της συνδρομής θα πρέπει να εφίστανται συνεχώς σεμινάρια, να παρακολουθούν συνεχώς σεμινάρια κατάρτισης και να ενημερώνονται για τις νέες μεθόδους. Και επίσης ήθελα να επισημάνω ότι η, Ευρωπαϊκή η Κροατία συγγνώμη, θέσπισε πολλά, πολλές νομοθετικές διατάξεις μετά, τη θέση ισχύ της, μετά την υπογραφή της ε, ενταξιακής συμφωνίας και εφόσον ε, τηρηθούν και πλήρως αυτές οι νέες νομοθετικές διατάξεις ε, θα θεσπιστεί στην Κροατία ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και η κανονικότητα των, της κοινοτικής χρηματοδότησης. Και η τελωνιακή έλεγχη στην Κροατία θα πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματική. Και θα πρέπει να γίνει καλύτερο ο συντονισμό μεταξύ των κονδυλίων που λαμβάνει η Κροατία από τα διαρθρωτικά ταμεία. Και καλό θα ήταν η χώρα αυτή να ιδρύσει ένα σύστημα προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τις άμεσες πληρωμές στη Γεωργία. Θα ήθελα να προσθέσω και δύο ακόμη τινά η Κροατία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής θέματα. Έχει συστήσει ένα νέο Υπουργείο για την κοινωνική χρηματοδότηση και μάλιστα ο αρμόδιος υπουργό θα είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάτι που συνιστά ένα πολύ χειρό μήνυμα εκ μέρους της Κροατίας. Επίσης έχει υιοθετηθεί ο νέος νόμος για τις ε, κρατικές προμήθειες και θα πρέπει φυσικά και αυτός να εφαρμοστεί πλήρως. Εν κατακλείδη λοιπόν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τα συμπεράσματα της ειδική έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Κροατία βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την ένταξη και θα είναι πλήρως έτοιμη για την ένταξη και για την ε, απορρόφηση Τη μεταξιακής χρηματοδότησης. Ευελπιστούμε φυσικά ότι θα τηρήσει και τι εκκρεμεί υποχρεώσεις της ε, η Κροατία πριν την οριστική της ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά την παρουσίαση και του εκπροσώπου του Ελεκτικού Συνεδρίου μπορούμε να συζητήσουμε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ja, vielen Dank, äh, Herr Berichterstatter. Bevor wir äh, den Vertreter σας ευχαριστώ. Τώρα θα ξανακούσουμε τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπενθυμίσω πως είχαμε ήδη τους ε, παρατηρητές από το Κροατικό Κοινοβούλιο και καλωσορίζω και τους παρατηρητές ε, στην Επιτροπή μας σήμερα νομίζω πως είναι πρώτη φορά καλώς ήρθατε λοιπόν κυρία Μαρινόβιτς, κυρία Πόσλαν Βράτ και Γεύκοβιτς ε, η Μπλέγκοβιτς ε, δεν τα είπα σωστά τα ονόματά σας, με συγχωρείτε τον Πρεντάν λοιπόν και τον Πρεντούσλη στην Επιτροπή μας Δίνω λοιπόν τον λόγο τώρα στον κύριο Φαζάκας ε, και μετά στους ε, δύο Πρώτα απ' όλα λοιπόν ο κύριος Φαζάκας από το Ελληνικό Συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν περάσω στα της έκθεσης να ευχαριστήσω εσάς και τον εισηγητή τον κύριο Τόμας Ντόιτς όχι μόνο για την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και επισήμως την έκθεσή μας αλλά για το ότι συζητάμε ξανά την ε, Κροατία ε, με βάση την ένταξή της και το ότι βεβαίω αποστελεί και εκπρόσωπο στο ελεγκτικό συνέδριο. Ίσως να είναι σύμπτωση ότι ασχολείται ένας ε, Ούγγρος ε, βουλευτής ε, και ο Ούγγρος ε, εκπρόσωπος του Ανακτικού Συνεδρίου. Γιατί εμείς ως γείτονας εδώ και 20 χρόνια καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια η Κροατία και η κυβέρνησή μας καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναγνωρίσει και την Κροατία όταν ανεξαρτοποιήθηκε και βεβαίως ε, σημαντικό ήταν πως ε, εντάχθηκε ως ε, συνδεδεμένο μέλος στην ΕΖΕΣ τότε η Κροατία και μην ξεχνάμε πως και άλλοι συνάδελφοι πριν από τέσσερα χρόνια άνοιξαν τον δρόμο της Κροατίας για την ένταξη. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον ε, εισηγητή αλλά βεβαίως και τους ε, προκατόχους μας εδώ πέρα για την πορεία της Κροατίας ε, την οποία προτίμασαν. Βεβαίως αυτή είναι μια πολιτική αξιολόγηση η οποία κανονικά δεν επιτρέπεται στο ελεγκτικό ε, συνέδριο, οπότε θα σας διαβάσω την εκθεσή μας στα αγγλικά όπως την έχω αποστείλει άλλωστε και στη γραμματεία για να περάσουμε στο επίσημο τμήμα της ε, παρουσίασής μας. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, κύριε συγητά, κύριε και κύριοι, πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη ε, τη δική μου για το ότι ετέθη η ειδική έκθεση στην ημερήσια διάταξη, η έκθεση για την ικανότητα της Κροατίας για να απορροφήσει τις ε, χρηματοδοτήσεις ε, μετά την ένταξη. Αναμένεται λοιπόν η ένταξη 1η Ιουλίου 2013 και έχει ήδη ξεκινήσει το 2001 η οικονομική βοήθεια στην Κροατία. Και οπωσδήποτε θεωρώ πως είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση. Το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε και τα συμπεράσματα της προηγούμενης ε, έκθεσης του που είχε σχέση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μεταξύ άλλων. Τότε έλεγε το ελεγκτικό συνέδριο πως οι δύο χώρες δεν είχαν την απαραίτητη ικανότητα να διαχειριστούν και να απορροφήσουν τα κονδύλια. Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτή την αξιολόγηση. Με την εμπειρία αυτή λοιπόν κατά νου, κατά τη σύνταξη της έκθεσης για την Κροατία επικεντρωθήκαμε στην διάσταση της δυνατότητας απορρόφησης της προενταξιακής βοήθειας. Εμείς δεν ελέγξαμε ούτε την ικανότητα γενικώ ένταξης της Κροατίας, ούτε ζητήματα διαφοράς. Όμως, όπως ανέφερε η πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την Κροατία ε, στις αρχές του έτους. Τα ζητήματα της ε, καταπολέμησης ε, της διαφθοράς στην Κροατία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Εάν τα μέλη της Επιτροπής σας θεωρούν αναγκαίο να συζητήσουμε αυτές τις στοιχές με περισσότερες λεπτομέρειες, το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να προετοιμάσει άλλη μία έκθεση σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ε, Κροατία. Ο έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου σκοπό είχε να απαντήσει το εξής ερώτημα. Ήταν αποτελεσματική η προενταξιακή βοήθεια στο να προετοιμαστεί η Κροατία στη διαχείριση των κονδυλίων. Επικεντρωθήκαμε σε δύο τομείς αξιολόγηση του εάν σχεδίασε η Επιτροπή τη βοήθεια της Ένωσης κατά τρόπον ώστε να βοηθάει ικανοποιητικά την Κροατία να προετοιμαστεί για τη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ένταξη και το εάν απέφεραν τα σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα όσον αφορά την ενίσχυση της ικανότητας Κροατίας να διαχειριστεί τα κονδύλια της Ένωση. Ο έλεγχο περιελάμβανε ανάλυση των εγγράφων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της πρωταξιακής βοήθειας, έλεγχο δείγματος 16 έργων τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ε, διαφορετικά μέσα σε συνεργασία με ε, υπαλλήλους της Επιτροπής και με τα Υπουργεία, Υπηρεσίες και Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές της Κροατίας. αξιολόγησή μας ήταν πως ε, συνεισφέρουμε στην αύξηση της διοικητικής ικανότητας της ε, Κροατίας, αλλά απαιτείται οπωσδήποτε περισσότερη ε, πρόοδος. Γεγονός είναι πως με την εισαγωγή το 2007 του ενιαίου μέσου του λεγόμενου μηχανισμού πρωταξιακής βοήθειας ε, έχει διευκολυνθεί κατά πολύ η διαδικασία και υπολογίσαμε πως υπήρξε μια αρκετά καλή διαχείριση των κονδυλίων χωρίς ελέγχους εξ άντε από πλευράς κομισιών όμως περισσότερο στο μης ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση διαρθρωτικών κονδυλίων και κονδυλίων συνοχής η Κομισιόν δεν έχει ακόμα εξουσιοδοτήσει την Κομισιόν να εφαρμόσει τέτοια βοήθεια χωρίς ελέγχους εκ των προτέρων γενικώ έχει ε, υπάρξει βοήθεια της Κομισιόν, την οποία περνούν και οι κροατικές αρχές. Όμως οι δυνατότητες δημοσίων προμηθειών ακόμη απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον επικεντρώθηκαν οι δυνατότητες αυτές και η παροχή αρχής στις κεντρικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές κατά κάποιον τρόπο παραμελήθηκαν παρά το ότι έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν στην εφαρμογή αυτής της χρηματοδότησης. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που επέτυχαν τα έργα αυτά, έχει υπάρξει σημαντική συνεισφορά στην οικοδόμηση της ικανότητας της Κροατίας για την διαχείριση της χρηματοδότησης μετά την ένταξη μέσω βεβαίως μιας μεθόδου πρακτικής εκμάθησης και υπάρχουν εδώ πέρα συγκεκριμένα παραδείγματα όπου έμεινε η εφαρμογή πολύ πίσω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Αυτό οφείλονταν σε καθυστερήσεις λόγω μη ε, οριμότητας των έργων όταν επιλέχθηκαν ή λόγω της έλλειψης, όπως είπα, δυνατότητας ε, διεξαγωγής δημοσίων προμηθειών. Επίσης, το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε πως υπήρχε ε, η τάση να υπάρχει επικέντρωση σε μεγάλα έργα και όχι σε μικρά ή μεσέ, τα οποία επίσης παίζουν σημαντικό ρόλο. Τέλος, λόγω των καθυστερήσεων και της έλλειψης έργων υπήρξε χαμηλή απορρόφηση ε, όσον αφορά τον τομέα της ε, αγροτικής ανάπτυξης. Οπότε το συνέδριο έκανε κάποιε συστάσει στι αρχέ τη Κροατία και στην Κομισιόν, όπου ορίζει του τομεί που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Συγκεκριμένα θεωρούμε πως θα πρέπει να αυξηθεί η προτεραιότητα που δίδεται στην δυνατότητα διεξαγωγής ε, διαγωνισμών δημοσίων προμηθειών για εκπαίδευση επιτόπου στην δουλειά και εκτός αυτής οικοδόμηση των δυνατοτήτων των περιφερειακών αρχών, ανάπτυξη των ε, δραστηριοτήτων που χρειάζεται για να υπάρξει πλήρης απορρόφηση της, ε, των διατίθεμων κονδυλίων και βεβαίως μέτρα καταπολέμησης της διαφοράς. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, κυρίες και κύριοι, βασιζόμενοι ε, στο ότι θα το επικυρώσουν τα κράτη-μέλη. Η Κροατία θα γίνει το 28ο κράτος μέλος σε 13 μήνες βεβαίως. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και οι αρχές της Κροατίας έχουν χρόνο να γίνει αυτό πριν από την ένταξη. Ταυτόχρονα η Κομισιόν πρέπει να λάβει υπόψη τα μαθήματα από την ένταξη της Κροατίας και να τα εφαρμόσει σε άλλες υποψήφιες χώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Φάζακας για αυτά τα οποία μας είπατε, εκπροσωπώντα το ελεγκτικό συνέδριο όσον αφορά την πολιτική αξιολόγηση της ε, κατάστασης ε, συμφωνώ και εγώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή όσον αφορά τώρα την περαιτέρω συζήτηση να σας πω πως πρέπει να ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 6 και 4 οπότε σας παρακαλώ να είστε σύντομοι και να ζητήσω από τις ε, συναδέλφους ε, της παρατηρήτριας από την ε, Κροατία να τους ρωτήσω ποιος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε παρά τις αρκετά θετικές αναφορές, την αρκετά θετική παρουσίαση. Γνωρίζουμε ότι μας απομένουν πολλές προσπάθειες και πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένε δράσεις και να σπίσουμε συγκεκριμένα μέτρα και να τα εφαρμόσουμε στο τομέα του δυναμικού απορροφήσεως σπόρων στην Κροατία. Θα ήθελα ιδιαίτερως να τονίσω κάποια βασικά σημεία που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά σήμερα. Πρώτα απ' όλα να τονίσω ότι όπως αναφέρεται και στην έκθεση, ότι συνδυάζοντας αρκετά θεσμικά όργανα που αναμειγνύονται στην διαχείριση των νέων πόρων στο νέο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Περιφερειακούς Πόρους του 2011, το Εκείνο 2011, δημιουργήθηκε αυτή, αυτός ο φορέας, τονίσαμε στην Κροατία πόσο σημαντική είναι η περιφερειακή ανάπτυξη το ότι ο ίδιος υπουργό διορίστηκε και σαν αντιπρόεδρος τη κυβερνήσεως, αυτό είναι κάτι που έστειλε ισχυρό πολιτικό μήνυμα και δείχνει πραγματική αφοσίωση της νέας κυβερνήσεω στα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης και της χρήσης των πόρων τη ευρωπαϊκή Ενώσεω. Αυτό το Υπουργείο στο μέλλον θα ασχολείται με τα ιδιωτικά ταμεία και θα παίζει το ρόλο ενό μη ενία διαχειριστική αρχή που θα ενισχύει το συντονισμό όλων των δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το πρώτο ήταν αυτό που ήθελα να τονίσω. Δεύτερον, σημασία έχει η αποδοτική χρήση των προενταξιακών μέσων, βλέποντας την αύξηση του δυναμικού τη Κροατίας για τη μελλοντική χρήση και απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής των Ιδιωτικών Ταμείων ήταν κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Γι' αυτό η διάθεση επαρκών δημοσιονομικών πόρων για την Κροατία είναι κάτι που σίγουρα θα συμβάλλει στη διαδικασία των οικονομικών μεταρρυθμίσεων που θα κάνει η Κροατία και κάτι άλλο που είναι σημαντικότατο είναι το περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφέρειες Κροατίας ανέπτυξαν το δυναμικό απορρόφησης για τους πόρους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι αρμοδιότητες τοπικής αυτοδίκησης των περιφερειών για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων έχει αξιολογηθεί επανειλημμένος και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν επαρκείς δυνατότητες. Παρ' όλα αυτά η Κροατία θα συνεχίσει την ενίσχυση των δομών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη της δρομολόγησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να βελτιωθεί το δυναμικό στο μέλλον. Και στο τέλος πρέπει να πω κάτι για τις ε, κρατικές προμήθειες. Τον Ιανουάριο του 2012 φέτος ψηφίστηκε νέος νόμος για τους ε, διαγωνισμούς ε, εξασφαλίστως διαφάνεια. Το 2011 χάρισε ένα πρόγραμμα ΥΠΑΡ που είχε τίτλο «Ενίσχυση του δυναμικού για τη κάλυψη, ε, διόρθωση ατασταλιών στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών» ήταν ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε χάρη στις πόσες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κατεβλήθησαν λοιπόν προσπάθεια για ευαισθητοποίηση για τα προβλήματα αυτά. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει η Κροατία την αύξηση του δυναμικού για τις κρατικές προμήθειες σε εθνικό αλλά κυρίως σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Λόγω όλων αυτών των προσπαθειών που θα αναλυθούν και στο μέλλον, πιστεύουμε ότι οι μελλοντικές εκθέσεις για την Κροατία θα είναι ακόμα καλύτερες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις δηλώσεις. Στην κυρία Μάκο να το τρώγω πρώτα. Ευχαριστώ, όπως είπε η συνάδελφος. Όπως και η συνάδελφος και εγώ θα είμαι πολύ σύντομη. Σε τοπικό επίπεδο βλέπουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η ανάπτυξη η περιφερειακή. Γιατί εκεί ζει κανείς την καθημερινή ζωή. πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Στις επικείμενες εκλογές οι πολίτες μας θα, θα κάνουν μια αποτίμηση του έργου της τοπικής αυτοδίκησης. Πόσον επιτυχώς απορρόφησαν τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Ομολογούμε ότι δεν ήμασταν πολύ καλοί όσον αφορά την απορρόφηση των προενταξιακών πόρων. Όμως, νομίζω ότι ήδη βλέπουμε να υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ τοπικών αρχών και αυτό υπόσχεται πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Πλένκοβιτς έχει το λόγο τελευταίος, εξού όμως. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω μερικά στοιχεία στα όσα είπαν οι συνάδελφοι και επειδή ήμουν πρώην ε, υπουργό για θέματα ε, ευρωπαϊκά, να τονίσω ότι η Κροατία τη δεκαετία του 90 δεν ήταν δικαιούχος προγραμμάτων βοηθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο για τεχνική ανάλυση του δυναμικού απορρόφησης την τελευταία δεκαετία. Διότι τα πρώτα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας διατέθησαν ήταν το FAR, το CARDS που ήρθαν μόνο στην προηγούμενη δεκαετία. Επιφέραμε πολλές βελτιώσεις όσον αφορά τη διαχείριση της βοήθειας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δημιουργήσαμε θεσμούς, φορείς και όπως αναφέρθηκε και στην έκθεση, πράττοντας μάθαμε, θεσπίσαμε ένα πλαίσιο που θα υπάρχει και μετά την ένταξη μετά που θα είμαστε πλήρη μέλη μετά την 1η Ιουλίου. Όπως είπε και πολύ σωστά ο συνάδελφος του ΕΛΚ, ο κύριος Ντόιτς, στην πρόταση ψηφίσματος ανέφερε κάποιες εκκρεμότητες. Αυτή η πρώτη ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ε, είναι λεπτομερής και αναλύει σωστά 16 προγράμματα που δειγματοδοτικά ελέγχθηκαν πέρσι είναι ένα καλό παράδειγμα για την γενική αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τη χρηματοδότηση στην Κροατία. Κάτι πιο θετικό. Προσθέτοντας τα όσα λένε τα δύο έγγραφα. Η Κροατία έχει υποβάλει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητά εξαίρεση από την αξιολόγηση εκ των προτέρων για καλύτερη σωστή οικονομική διαχείριση και καλύτερο έλεγχο της χρήσεως των πόρων και των προγραμμάτων και πώς υλοποιούνται τα προγράμματα. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν τα στοιχεία για να προετοιμαστεί η Κροατία ούτω ώστε να έχει πιο όρημα προγράμματα στο χαρτοφυλάκιό της για να αυξήσει το δυναμικό απορρόφησης από τη στιγμή θα γίνουμε μέλη και από τη στιγμή που θα τίθενται τα διαθωτικά ταμεία, η πόροι των διαθωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κροατία θα χρησιμοποιήσουν αυτό, αυτή τη χρονιά, κυρίω με το τροποποιημένο σύστημα που ανέφερε η κυρία Βέρμπατ, με το νέο Υπουργείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, που θα διαχειρίζεται στου πόρου. Και κάτι λιγότερο από 13 μήνες που μας περιμένουν είναι πολύ σημαντική για την επιτυχή ε, εκτέλεση του έργου που έχουμε αναλάβει. Ευχαριστώ για τη συνεργασία που έλαβε χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο. Ε, θα ήθελα πρώτα να υπογραμμίσω μάλλον ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ θετική. Το ότι έχουμε δηλαδή ε, συμμετοχή των παρατηρητών σε αυτή την πρώιμη φάση της συζήτησης και πριν την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έτσι έχουμε και τις δικές σας ε, απόψεις και τα σχόλιά σας για το θέμα, αλλά και στο Ζάγκρεπ θα έχουμε ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με τη Βέσνα Πούσιτς, την Υπουργό Εξωτερικό σας. Και επίσης προσβλέπουμε σε πιο τακτικές ανταλλαγές απόψεων όσο προχωρούμε ε, και πλησιάζουμε πιο κοντά στην επίσημη ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα ήθελα να δώσω τη δυνατότητα και στην Κομισιόν να τοποθετηθεί. Καλωσορίζω τον κύριο Ντύρ Κλάγκε από την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης ε, Τμήματάρχης. Ε, εάν ε, θέλετε το λόγο τον έχετε. Ευχαριστώ, θα είμαι εξαιρετικά λακωνικός. Θα ήθελα να πω ότι γενικώ επιδοκιμάζουμε την αξιολόγηση του ελεκτικού συνεδρίου και παρακολουθούμε και εμείς μαζί με την Κροασία, μαζί με την Κροατία την προσπάθεια υιοθέτηση των συστάσεων και της εφαρμογής των συστάσεων του ελεκτικού συνεδρίου. Αναφέρθηκαν κάποια προγράμματα ανάπτυξη πέθρου. Ήδη τροποποιήθηκε το σχετικό πρόγραμμα ανάπτυξη πέθρου προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία για τι δημόσιε προμήθειε. Ήδη από τις αρχές του έτους ισχύει η νέα νομοθεσία για τις κρατικές προμήθειες. Ε, ευελπιστούμε ότι θα εφαρμοστεί πιστά. Σε ό,τι αφορά τα όρημα σχέδια, το θέμα αυτό είναι ένα ε, θέμα που αναφέρθηκε πολλές φορές και υπάρχει το πρόγραμμα Γιάσπαρ για την προώθηση τέτοιων προγραμμάτων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες προκειμένου να δημιουργηθούν ε, όρημα προγράμματα και να υποβληθούν όρημα σχέδια και μάλιστα η σχετική απόφαση ελήφθη το Μάρτιο φέτος. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των τοπικών και περιφερειακών αρχών και ε, παρέχεται συνδρομή και για τις διάφορες συνιστώσεις αυτής της ανάπτυξης της διοικητικής ικανότητας. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε είναι η συνέχιση της χρηματοοικονομικής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Μάλιστα είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στο θέμα αυτό, στα πλαίσια του ΙΠΑ, της προτεξιακής συνδρομής, προκειμένου να παταχθεί η διαφθορά. Σε ό,τι αφορά τον εξάντε έλεγχο, τον πρόωρο έλεγχο που θα πρέπει το αργότερο να γίνεται μέχρι την ένταξη της χώρας για τις συνιστώσεις 4 και 3 και 4, έχουμε στενή συνεργασία με τους Κροάτες συναδέλφους Στόχο μας είναι η εξαίρεση αυτή να υλοποιηθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου, δηλαδή μισό, χρόνο, μισό έτος, ένα εξάμεινο πριν την ένταξη. Θα συνεχίσουμε πάντως την στενή συνεργασία με την Κροατία προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή της προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθιστώντας, καθιστώντας τη χώρα καλά προετοιμασμένη για να αξιοποιήσει την μετενταξιακή χρηματοδότηση. Αναφέρθηκε και η έκθεση παρακολούθησης που δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο η Κροατία. Η επόμενη περιεκτική έκθεση ελέγχου και παρακολούθησης θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο. Θα την ε, παρουσιάσουμε φυσικά και στα κρατημέλη και θα είναι και ένα οδηγό για την Κροατία για να συνεχίσει την εφαρμογή και τι προετοιμασίε για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλος, τον λόγο έχει ο κύριος Σίγητης. Έχει τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να είμαι Να πω κάποια πράγματα για αυτά τα οποία ακούστηκαν. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι βρίσκονται εδώ Κροατοί παρατηρητές, οι Κροατοί παρατηρητές μας και, και συμμετέχουν σε αυτό το δημοκρατικό πνεύμα, έτσι είναι πιο δημοκρατική όλη η διαδικασία. Είναι λοιπόν ευπρόσδεκτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αποφασίσει σε ζητήματα που αφορούν την Κροατία χωρίς τη συμμετοχή των ε, Κροατών συναδέλφων. Οι κροατικές αρχές οπωσδήποτε θα πρέπει να εργαστούν σκληρά τους επόμενους 13 ε, ε, μήνες. Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά τα οποία ακούσαμε από την Κομισιόν. Οι όροι ένταξης είναι πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουν να είναι αυστηροί στο μέλλον, αλλά νομίζω πως οι αρχές της Κροατίας ε, έχουν ε, αποδειχθεί ικανές ε, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν κράτη-μέλη εντό της Ένωσης τα οποία παρά το ότι είχαν την δυνατότητα συμμετοχής ε, και χρηματοδότησης ε, είναι σε ένα βαθμό κανονικότητας ε, των έργων τους που δεν είναι θα έλεγα η βέλτιστη σε σχέση μάλιστα και σε σύγκριση με την Κροατία οπότε νομίζω πως είναι ικανοποιητικό το 2015 ή 2014 όταν θα εξολογήσουμε την απόδοση της ε, Κροατίας ε, καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ε, η απόδοση της Κροατίας ή δηλαδή το ποσοστό απορρόφησης ή η ποιότητα των έργων είναι εξίσου καλή με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο και έχουμε κάθε λόγο να το πιστεύουμε αυτό με βάση την έκθεση του Ελληνικτικού συνεδρίου. Να επαναλάβω δε αυτό το οποίο είπα στην πρώτη μου παρέμβαση. Εγώ είμαι πεπισμένος πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ισχυροποιηθεί με την ένταξη της Κροατίας. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας για αυτά τα οποία μας είπε στο τέλος με τα οποία μπορώ να συμφωνήσω και εγώ θεωρώ πως είναι θετικό και δημοκρατικό το ότι βρίσκονται εδώ οι παρατηρητές. Φτάσαμε λοιπόν στην ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών που είναι 8 Ιουνίου, 12 η ώρα και ευχαριστώ και τον κύριο Φάζακας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον κύριο Λάγκε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, αλλά και τη γραμματεία, τους διερμηνείς και φτάσαμε νομίζω στο τέλος της ε, συνεδρίασης. Η επόμενη συνεδρίαση ε, έχει ήδη προγραμματιστεί.